Ε, Καλησπέρα σας. Παρακαλώ καθίστε. Θα ξεκινήσουμε την ψηφοφορία εντός ολίγου. Απλώς προηγουμένως να δώσω το λόγο στην κυρία Κοράτσα Μπίλτ που τον ζήτησε. Thank you, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να σας ε, ρωτήσω. Η έρευνα του Κοινοβουλίου για την απάτη ε, με την